επίση τον ε, Επίτροπο κύριο Ναύρα, που εκπροσωπεί την υπάτη πρόσωπο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Το Σώμα ενέκρινε μια σειρά από ψηφίσματα για την κατάσταση στη δημοκρατική, στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και πιο συγκεκριμένα για την κατάσταση στις ανατολικές ε, μεθοριακές περιοχέ. συμπεριλαμβανομένων και του Κιβού. Γνωρίζετε την ε, απαράδεκτη βία που σημειώνεται από το περασμένο φθινόπωρο, ιδιαίτερα στο βόρειο Κιβού. Ορισμένες ε, περιοχές έχουν θυγεί πολύ άσχημα. Οι νεκροί στην ε, περιοχή των Μπένι εκτιμούνται από την κοινωνία των πολιτών σε 550 από το Σεπτέμβριο του 2014. Επιπλέον, δεκάδες χιλιάδες κατοίκων έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά. Φυσικά, η πρώτη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ανθρωπιστική πρόσβαση και καλούμε για άλλη μια φορά να σταματήσει η προσπάθεια να απαχθούν στοχευμένα οι εργαζόμενοι για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι πράξεις αυτές είναι σύμφωνες με τον κανονισμό 1257 κάθετος 96, ιδιαίτερα ε, γιατί οι ενέργειες των ε, συνεργατών μας γίνονται με βάση την αρχή της μη διάκριση. Οι ενέργειες βίας συνεχίζονται γιατί δεν υπάρχει καμία κρατική παρουσία. Οι υπηρεσίε και οι θεσμοί που θα έπρεπε να προλάβουν τη βία και να τη σταματήσουν και να αναλάβουν νομική δράση κατά των υπετίων απουσιάζουν, δυστυχώ. Η προσπάθεια δημιουργία κρατικών θεσμών στη χώρα αυτή εμποδίζονται από την παρούσα αβεβαιότητα για το πότε θα διεξαχθούν εκλογές που με βάση το Σύνταγμα θα πρέπει να διεξαχθούν φέτος. Μία άλλη πλευρά που συνεχίζει να παίζει ρόλο είναι, είναι η εκμετάλλευση από πολλέ πλευρέ και των ε, αγρίων ζώων και διαφόρων φυσικών πόρων. Μια πρόσφατη έκθεση μιας ε, ομάδας συμπρογνωμόνων του ΟΗΕ τονίζει ότι συνεχίζει να συμμετέχει η οργάνωση Lord's Resistance Army. Συμμετέχει σε λαθροθυρία και συνεχίζει να γίνεται εξόριξη χρυσού, η οποία, ο οποίος χρυσό μετά περνάει στη διεθνή αγορά. Κάπως μας παρεχωρεί το γεγονός ότι ορισμένες ένοπλες ομάδες έχουν λιγότερες ευκαιρίες να ωφεληθούν από αυτή την παράνομη συμμετοχή τους στην εξόρυξη του ταντάλιου, του τουμστενίου και του κασιτέρου λόγω των προσπαθειών που γίνεται για να έχουμε συστήματα ανιχνευσιμότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει τις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει τη διάσταση με πρώτων υλών και φυσικών πόρων αυτής της προσπάθειας. Καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντική η αντιμετώπιση των βασικών αιτίων αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί που κάνουν αυτές τις πράξεις έχουν δικαιολογία. Αυτό έχει να κάνει και σε αυτούς που παροτρύνουν σε βία και που στέλνουν μηνύματα μίσους. Ορισμένα άτομα και όχι κοινότητε και εθνοτικέ ομάδε είναι πέντε για αυτέ τι ενέργειες. Όπως επανειλημμένα έχει υποθεί και εδώ στο σώμα, οι δραστηριότητε αυτών των ενόπλων ομάδων στην ε, ανατολική περιοχή της χώρα αυτής είναι προσβολή για τους πολίτε. Υπονομεύει και τα ανθρώπινα και τα νομότυπα δικαιώματά τους. Καταστρέφει την ειρήνη και καθιστά πολύ δύσκολο να προγραμματίσει κανείς τη ζωή του και να σκεφτεί για το μέλλον. Για να σταματήσουν να δρούν οι ένοπλες ομάδες χρειάζεται ένα ουσιαστικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των όπλων δυνάμεων της χώρας και του Μονούσκο. Και πρέπει να υπάρξει αυτή η συνεργασία σύντομα. Η συμφωνία με της αρχής ήδη επετέφθη το Φεβρουάριο, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί. Και επίση, ε, η επιβολή τη δικαιοσύνη είναι σημαντική. Πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση και της πολιτικής και της στρατιωτικής δικαιοσύνη. Και επιμένουμε ότι όσοι βοηθούν ή συνομωτούν με τις ένοπλες ομάδες πρέπει να διωχθούν. Οι σοβαρέ ε, φρικαλότες που έχουν ε, λάβει χώρα στα ανατολικά της χώρας πρέπει να διερευνηθούν και να διωχθούν οι κυρίως υπεύθυνοι για να διερευνήσουν και να ε, διώξουν τους υπέτειους είναι οι αρχές της χώρας όπου ε, έλαβαν χώρα αυτές οι ενέργειες η χώρα των οποίων είναι πολίτες. Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε τη χώρα για να δημιουργηθούν οι δομές και να βοηθηθούν από ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο για να καθιστούν εφικτά όλα αυτά. Κύριε Πρόεδρε, να στραφώ τώρα στο ευρύτερο αλλά κρίσιμο ε, ζήτημα της διακυβέρνησης επίκυνται εκλογές σε μερικούς μήνες. Η χώρα λοιπόν είναι σε ένα κρίσιμο σταύρο δρόμο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας μέσω της αποφάσεως 2277, του ψηφίσματος 2277, ε, έθεσε ε, την αφετηρία αυτής της διαδικασίας. Αυτό το ψήφισμα εγκρίθηκε τον ε, Μάρτιο και τονίζει ότι είναι ευθύνη των αρχών της χώρας να διεξαγάγουν εκλογές με βάση τις διατάξεις του συντάγματος. Φυσικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει ότι η απόφαση του Σταματικού Δικαστηρίου της χώρας το Μάιο τρέχοντος παίζει το ρόλο της και σεβόμεθα την κυριαρχία της χώρας. Παράλληλα και στα πλαίσια όχι μόνο της Συμφωνίας Κοτονού αλλά και της ε, Χάρτας Δημοκρατίας Εκλογών και Διακυβέρνησης της, του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας τονίζουμε ότι μια δημοκρατική κυβέρνηση δημιουργεί την νομοποίησή της ε, με βάση τακτικέ εκλογέ με βάση τις προθεσμίε του συντάγματο. Για να υπάρξει συνένεση που να οδηγεί σε εκλογές χρειάζεται πολιτικό διάλογο. Επιγόντω. και ταχαίω, ο διάλογο πρέπει να είναι στοχευμένο. Όλε οι αντιπροσωπευτικέ πολιτικέ δυνάμεις πρέπει να συμμετάσχουν. Ένα τέτοιο διάλογο θα πρέπει να έχει ω κύριο στόχο ένα σαφή οδικό χάρτη που να έχει και χρονοδιάγραμμα και πρόγραμμα χρηματοδότησης ούτως ώστε να γίνουν ούτω ώστε να γίνουν νομότυπε εκλογέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη, τον Οργανισμό Αφρικανική Ενότητα και την OIF επανέλαβαν στι 6 Ιουνίου τη σημασία του ε, Χάιντεμ Κότσο και της αποστολής που έχει αναλάβει υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλήγοντας, θεωρώ ότι οι επιτυχείς εκλογές θα εξαρτητούν όχι μόνο από την αναγκαία τεχνική υποδομή, αλλά από την επίτευξη του αναγκαίου κλίματος σεβασμού των δικαιωμάτων και ελευθεριών, του δικαιώματος ελευθερίας έκφρασης και του συνέρχεστε. Ούτω ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πολιτικού διαλόγου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Επιτροπή για το των πολιτικών ομάδων. Πρώτα πρώτα κυρία Μαρία Γκάμπριελ για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε επίτροπε. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξεκινήσω μιλώντας για τον ε, εκδημοκρατισμό, το δημοκρατικό προτσέζ για τη Δημοκρατία του Κόγκορα. Ε, μου έρχεται το, το, το ευμετάβολο, μου έρχεται το, το ευάλωτο στο μυαλό. Αυτό είναι το θέμα της ε, ευθύνη μα. Οπότε μιλούμε για τι σφαγέ αυτέ στο Ανατολικό Κονγκό, αλλά περίπου όλα αυτά να τα δούμε στο ευρύτερο πλαίσιο και γι' αυτό θέλω να σταθώ στα εξή τρία σημεία. Πρώτα-πρώτα, θα πρέπει να πέσει άπλετο φω όσον αφορά αυτέ τι σφαγέ των Ανατολικών με τη χώρα. Θα πρέπει να σταθούμε τη δικαιοσύνη υπεύθυνη και θα πρέπει η συνεργασία να συνεχιστεί μεταξύ τη Μόνουσκο και των ενόπλων δυνάμεων και να υπάρχει μια διευρυμένη εντολή. Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να καταπολεμεί την ατιμορρησία, θα πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση ε, και να φέρει αποτελέσματα η προσπάθεια ε, στον τομέα της δικαιοσύνης και της ασφάλειας. Τώρα όσον αφορά την εκλογική διαδικασία θα πρέπει να προσέξουμε ότι τα προβλήματα στον τομέα της ε, ασφάλειας να μην υπονομεύσουν και τις ε, εκλογές που θα πρέπει να διεξαχθούν. Ούτε οι εκλογές αντίστοιχα να επηρεάσουν την ασφάλεια. Γιατί είδαμε τι έγινε μετά τις εκλογές του 2011. Όλα έχουν σημασία και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να υπάρχει ζωντανό διάλογος μεταξύ ε, των δύο πλευρών. Και οπότε δεν θα πρέπει να παραβλάψουμε την κοινωνία των ε, πολιτών, γιατί συνήθως αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει μπλοκάρισμα στις πολιτικές εξελίξεις. Ε, οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνουν οι εκλογές, τι θα γίνει με τους νέους, ε, με τα δημοσιονομικά και οπότε μπορούμε να διαμαζούμε σημαντικό ρόλο και ε, μην είμαστε απλώς διαμεσολαβητές. Θα πρέπει εμείς και η διεθνής κοινότητα ήδη έχουμε πει να, να ότι είμαστε δημοσιολαβητές αλλά πρέπει τώρα να είμαστε πιο δυναμικοί και θα πρέπει να ρίξουμε το δικό μας βάρος γιατί θα πρέπει να δούμε ότι όλους τους χρειάζεται σε διαδικασία της Αντισαβέμπα ή η Αφρική και να υπάρξει ασφάλεια και ειρήνη στις μεγάλες λίμνες. Οπότε χρειάζεται ένα συντονισμός να τηρηθεί το ισχύον σύνταγμα ούτω ώστε να μην πέσουμε σε κάποια ε, κλίμακα ε, τεράστια σε ανθρωπιστική κρίση. Τώρα, για τους σοσιαλδημοκράτες ο Πρόεδρος Πιτέλα. Κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να σας ομολογήσω ότι πολλές φορές αισθάνομαι ότι λέμε τα ίδια αυτούς τους εμπειρογνώμονες. Ε, αυτό ε, κάτι το οποίο μου φέρνει ανατριχίλα γιατί όντως το σοβεί μια σύγκρουση αλλά πρόκειται για μια σύγκρουση λένε χαμηλής έντασης, χαμηλής έντασης, μα τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε 6 εκατομμύρια νεκρούς, 1,5 εκατομμύριο ε, από εκτοπισμένους. Οπότε αν κάνετε αυτόν τον... Ε, ε, θα έχουμε 300.000 νεκρούς το έτος 8.000 την ημέρα και λέμε για χαμηλές ένταση σύγκρουση. Εγώ νομίζω ότι αντί γι' αυτό θα πρέπει να λέμε ότι πρόκειται για σύγκρουση πολύ χαμηλής προσοχής, προσοχής που της δίνει η διεθνής κοινότητα σε αυτή την ε, τραγωδία που έχει κάποιες ε, τρομακτικές διαστάσεις και γι' αυτό σας λέω ότι σήμερα εμείς θέλουμε να στραφούμε πάνω απ' όλα στην υπάτη εκπρόσωπο Φεντερίνα Μογκερίνη. Θα πρέπει να επιδείξουμε ευαισθησία γιατί θα πρέπει από κοινού να σταματήσουμε την κλιμάκωση της βίας εις βάρος ε, αυτού του απροστάτευτου ε, πληθυσμού από ε, τους παραστατιωτικούς οι οποίοι θέλουν να ελέγξουν αυτή την περιοχή που είναι από τις πιο όλο τον κόσμο όσον αφορά τους φυσικούς πόρους και τα, τα ορυκτά. Είναι ξεκάθαρο το ότι πρέπει να κάνουμε πρώτα-πρώτα. Θα πρέπει να υπάρξει συγκρότηση ανεξάρτητης Ελληνικής Επιτροπής διεθνούς επίπεδου και θα πρέπει να ρίξει άπλετο φως στις ε, αιτίες αλλά και στους ε, υπεύθυνους αυτής της σφαγής. Δεύτερον, θα πρέπει να ζητήσουμε να εμπλακεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ε, όσον αφορά όλα αυτά το πήγαιναν στο Μπένι. Επίση, θα πρέπει να ζητηθεί μια έκθεση αξιολόγηση του ΟΗΕ όσον αφορά τα αποτελέσματα τη αποστολή Μονούσκο και επίση θα πρέπει να υπάρξουν δυνάμει του ΟΗΕ και επιτόπου να έχουν ε, την εντολή της παρέμβασης για την προστασία του ναμάχων. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητηθεί και να απαιτηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ό,τι μπορεί και αυτό να να οδηγήσει στην, στο σταμάτημα αυτή τη σύγκρουση. Οπότε εμεί ω δημοκράτε, δημοκράτες θα στείλουμε στο Κύβο την ε, συνάδελφο Ελένα Βαλεντιάνο που είναι πρόεδρο τη ε, Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να συναντηθεί με του παράγοντε τη κοινωνία πολιτών τη ε, χώρα και των άλλων προσώπων του λαού επιτόπου. Και όταν γυρίσει θα συζητήσουμε όλα αυτά με όλου του συναδέλφους του Κοινοβουλίου, με όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης και φυσικά με το Προεδρείο μας και με την είπατε εκπρόσωπο κυρία Μογκερίνη. Θα πρέπει να ξυπνήσει η διεθνής κοινότητα. Wake up, μην εγκαταλείπετε στην τύχη τους τους ε, Κογκολέζους του Κίβου. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η βία που εδώ και 20 χρόνια αυξάνεται χωρίς σταματημό. για το ECR τώρα. Κύριο Μάκερα. Ευχαριστώ. Το Κόγκο είναι ο τόπος, το σημείο της μεγαλύτερης τραγωδίας στην οικουμένη και <clears throat> κάποιος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ε, τα πράγματα αποκαλεί τη σπασμένη καρδιά της Αφρικής στο Κόγκο και πολύ λίγη προσοχή στρέφουμε στο Κόγκο και ουσιαστικά πρόκειται για μια λαιλασία που παραμένει αναλύωτη και ε, βλέπουμε ότι στο Ανατολικό Κονγκό σφαγιάζονται άτομα με μαχαίρια, με ματσέτες, ε, βιάζονται γυναίκες και κορίτσια και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Πρόκειται για τη διασφάλιση της εξουσίας από πλευράς Προέδρου Συζητώντα πριν από μήνε για την κατάσταση την ανθρωπιστική στον Κονγκό, τα αναφέραμε αυτά, δεν υπήρξε όμω καμία πρόοδο από τότε. Το αντίθετο, είχαμε την ε, ε, δίκη κατά του ε, Κατούμπη, ωστόσο η κρίση επιδεινωνόταν και επεκτηνόταν επί τόπου. Πρέπει κάθε μέσω να χρησιμοποιήσουμε ώστε να αποφευθεί ένας νέος ε, αιματηρός εμφύλιος πόλεμος. Δεν πρέπει να διατηρηθεί αυτή η περιφερειακή διάσταση σε αυτόν τον πόλεμο. Πρόκειται όμως για πρώτες ύλες και η μεγαλύτερη κατάρα του Κονγκό είναι ο πλούτος του σε αυτούς τους φυσικούς πόρους σε αυτές τις πρώτες ύλε. Πρέπει να αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το εμπόριο ορυκτών και μετάλλων είναι ένα από τα αίτια αυτής της κατάστασης. Εκείνοι που επιθυμούν να εισαγάγουν αυτά τα ορυκτά και μέταλλα πρέπει να αποδεικνύουν ότι δεν αποτελεί αυτό συνεισφορά στην βία και συμμετοχή στις βιοπραγίες θα πρέπει η Μινούσκο η Αποστολή Ηνωμένων Εθνών και πρέπει με κάθε τρόπο να προσπαθήσουμε να εξουδετερώσουμε αυτή την κατάσταση. Κύριος Γκέρενς, με αυτό το ψήφισμα λέμε ότι θα πρέπει να κάνουμε τη διαφορά, να σταματήσει αυτή η τραγωδία που γίνεται στο βορειοανατολικό Κονγκό. Προσφοράψαμε πέντε πολιτικές ομάδες. Διπλωματία θέλουμε, υπεύθυνη πολιτική, ούτω ώστε να σταματήσει αυτό ο βαρβαρισμός που μαστίζει την ζωή των αμάχων παιδιών, ε, γυναικών και χθε στην Χάγη έκρινε για την Πέμπα ε, το Διεθνές Δικαστήριο και είπε ότι θα πρέπει να υπάρξουν αποδείξεις και να να ενώπιον της δικαιοσύνης οι αληθείς υπεύθυνοι για αυτή την ε, σφαγή. Οπότε και το Συμβουλίο Ασφαλείας θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτά τα γεγονότα. Ό,τι γίνεται ακόμα στο Βόρειο Κύβο και να δούμε σε ποιο βαθμό η Μονούσκο μπορεί να βοηθήσει ούτω ώστε πάλι να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα θεμελιώδη. Ολοένα γιατί η κατάσταση επιδεινώνεται στο Κονγκό και οπότε έχουμε βέβαια τις ε, επιχειρήσεις που ωφελούνται από τους φυσικούς πόρους της ε, χώρας οπότε μόνο έτσι ε, αν το δούμε μπορούμε κάτι να κάνουμε κατά του οργανωμένου εγκλήματος και να μπορέσουμε ιδίω στο βορειακή αυτούς τους να τους ε, αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει επίσης ε, να δούμε τι λένε, τι θέλουν οι οι Αφρικανοί και αυτοί να μας δώσουν ε, την καθοδήγηση για το τι θα κάνουμε για να σταματήσει το φαινόμενο. Και τώρα, για την Συνομοσπονδιακή Αριστερά έχει τον λόγο η κυρία Ροντρίγκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να τοποθετηθούμε για να καταγγείλουμε την κατάσταση στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αυτή τη φορά η κατα... καταγγελία και καταδίκη μας σε σχέση με τις σφαγές στο Ανατολικό Κονγκό με τις, ε, την επίλυση την ειρηνική του, της σύραξης ε, πρέπει να προχωρήσουμε. Οι στρατιωτικές λύσεις συνεπάγουν μεγαλύτερη βία και δεινά για τον πληθυσμό εκφράζουμε την ανησυχία μας για την ενίσχυση της στρατιωτικής εντολής και παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αφρική και τον ρόλο του σε διάφορες χώρες καθώς και στην λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Ζητούμε την διάλυση και την απόσυρση του Αφρικόμ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξεκινήσει μια ανεξάρτητη εξέταση για το ρόλο των ευρωπαϊκών πολυεθνικών όσον αφορά την παραβίαση κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και των δεσμών τους με την χρηματοδότηση ένοπλων ομάδων και συμμοριών για να μπορούν να ε, συνεχίσουν να λαιλατούν την επικράτεια του Κονγκό. <clears throat> Θα πρέπει σε σχέση με τα όσα αποφασίστηκαν το 2015 για το περιβάλλον, όπου αναφέρθηκε ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό της εκ των φυσικών πόρων χρηματοδοτούσαν ακριβώς αυτέ τι ένοπλες συμμορίες. Να το λάβουμε υπόψη επίση πρέπει να εγγυηθούμε την μη ανάμειξη και το σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων τη ανεξάρτητης Λαική Δημοκρατία του Κονγκό. Να σεβαστούμε αυτή την πολιτική κυριαρχία, κυριαρχικά δικαιώματα σημαίνει ότι θα πρέπει να μπορούν να υποφεληθούν οι Κονγκολέζοι από τον φυσικό του πλούτο. Γι' αυτό πρέπει να αποκατασταθεί ο έλεγχο ε, στι δραστηριότητε των πολιεθνικών μέσω την ακύρωση και οποιονδήποτε συμβάσεων ε, ε, για την εκμετάλλευση ορυκτών, μετάλλων ε, ή των τροπικών δασών. Επίσης η αντιμετώπιση της υπερχρέωσης του χρέους πρέπει να αναλυθούν τα αναγκαία μέτρα για να ανταποκριθούμε στις πιο βασικές ανάγκες του πληθυσμού του Κονγκό. Ευχαριστώ. Για τους Ευχαριστώ. Και σήμερα, για άλλη μια φορά, καταδικάζουμε την τρομερή κατάσταση στο Κονγκό, ιδιαίτερα τις ε, σφαγές που γίνονται στα Ανατολικά. Θα καταλάβετε, κύριε εκπρόσωπο τη Κομισιόν, ότι είμαστε ιδιαίτερα απογοητευμένοι, γιατί πριν από λίγο χρονικό διάστημα είχαμε κρίνει μία άλλη και δεν βλέπουμε να έχει καμία επίπτωση στην κατάσταση επιτόπου, στην τρομερή κατάσταση που ζει ένα μεγάλο τμήμα το πληθυσμό. Χαιρόμαστε για αυτό το κοινό ψήφισμα. Ένα ψήφισμα την οποία υπογράφουμε Υπάρχει συνένεση, αλλά θα θέλαμε να είναι πιο κατηγορηματική σε ορισμένα σημεία, ιδιαίτερα όταν ε, κρίνουμε το ρόλο της Μονούσκο, της ε, αποστολής σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κονγκό. Γιατί ορισμένοι ανεξάρτητοι παρατηρητές ε, τη θεωρούν παθητική, αδρανή. Δεν, κάνει τον, δεν παίζει το ρόλο της να, να προστατεύσει δηλαδή, τον πληθυσμό από αυτές τις φαγές. Επίσης ε, ελπίζουμε η έρευνα που ζητάμε να διεξαχθεί για να δούμε ποιο είναι υπεύθυνο εάν δεν εκτελεί τα καθήκοντά τη ε, Χαιρόμαστε που αναφέρονται κάποια σημεία για το πόσο τρομερή είναι η κατάσταση στο Κονγκό. Πρώτον, το ότι οι γυναίκες είναι το θύμα, τα θύματα ε, και ότι βιάζονται ε, γυναίκες και κορίτσια και στρατολογούνται ε, στρατιώτες, μαχητές, παιδιά που δεν έχουν μετά καμία δυνατότητα να έχουν μια κανονική ζωή και επίσης ότι εκμεταλλεύονται τα ορεικτά. Και εδώ η Κομισιόν πολλά μπορεί να κάνει γιατί παίζουν ρόλο ευρωπαϊκέ εταιρείε. και πρέπει να ξεπεράσουμε τι απλέ διακηρύξεις. Πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα κυρώσεων ερευνών για να δούμε ποιε ευρωπαϊκές πολυεθνικές συμμετέχουν σε αυτό το εμπόριο. Γιατί αυτό είναι σε τελευταία ανάλυση ο λόγο για την τρομερή κατάσταση στην περιοχή αυτή. Ένα θέμα του ψηφίσματος αναφέρει τη δυνατότητα κυρώσεων για αυτούς που είναι άμεσα υπέτη για αυτές τις ε, σφαγέ. Να μην μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια, να καταδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εγκαταλείπει τον πληθυσμό του Κονγκό. Ευχαριστώ πολύ. Για την ομάδα Ευρώπη της Ελευθερίας και της Άμεσης Δημοκρατίας, ο κύριος Κοράου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από το 1960 έχουμε στο Κονγκό αυτή την ε, βία που συνεχίζεται και κορυφώθηκε τα τελευταία χρόνια. Ο πρόεδρος Καμπίλα ε, δεν φροντίζει το πώς θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Το μόνο που θέλει είναι πώς θα κρατηθεί στην εξουσία για να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Το είπαν πολλοί συνάδελφοι. Είναι τραγική στις ανατολικές περιοχές, στο Κιβού και στην Κατάγκα η κατάσταση και πάντα για τον ίδιο λόγο ο πλούτος της χώρας, η εκμετάλλευση των πόρων, των πρώτων υλών, των ε, ορυκτών γεμετάλλων. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε πιο αυστηροί σε σχέση με τις πολυεθνικές, τις ευρωπαϊκές που βρουν στην περιοχή. Θα πρέπει επίσης να γίνει κάποια ανεξάρτητη έρευνα ε, ε, χέρι-χέρι με την αποστολή την Μονούσκο. Ε, γιατί έχουμε τώρα τη δυσκολία του να κατέβουμε σε κάποια συμπεράσματα για αυτή την έρευνα και είδαμε ότι τελικά δεν προέκυψε τίποτα όσον αφορά ε, την εξόριξη, όσον αφορά τα ορυκτά και το εμπόριό τους. Οπότε νομίζω ότι κάνουμε τόσο πολλά τόσο χρόνο, αλλά ήρθε η ώρα να πετύχουμε κάτι συγκεκριμένο. Ιδάλλως θα μιλάμε και θα μιλάμε ε, χωρίς να πετυχαίνουμε τίποτα. Γιατί το ο ευχαριστήσω και δεν το κάνω συχνά τους συναδέλφους για το σωστό τρόπο που αναλύνει την κατάσταση στο, στο Κονγκό, την, ε, ιδιαίτερα τον κύριο Πιτέλα. Αγαπώ πολύ αυτή τη χώρα. Ήμουν ε, κοντά στον αντιπρόεδρο Ζαντίν Γκομά κατά την περίοδο μετάβαση και συμμετείχα σε αυτή τη μετάβαση. Οι δυσκολίε ε, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκύπτουν από τα πλούτη τη χώρα. Υπενθυμίζω ότι ο Λοράν Ντεζιρέ Καμπιλά επελέγει γιατί η Ουγγάντα και η Ρουάντα είχαν αποφασίσει με εντολή μια εξωτερική δύναμη και μπορώ να σα πω ποια ήταν αυτή η εξωτερική δύναμη, αν θέλετε, να εισβάλλουν στη χώρα. Και ενώ ο Λοράν Ντεζιρέ Καμπίλα ε, εισέβαλε στη χώρα, ορισμένε επιχειρήσει υπέγραφαν συμβάσει αμερικανικέ. Και όταν ο Λοράν Ντεζιρέ Καμπίλα ε, άλλαξε στάση και αποφάσισε να στηρίξει τα συμφέροντα της ε, χώρας του αποφασίστηκαν αποφασίστηκε εδώ στις Βρυξέλλες και ξέρω ποιοι ήταν και με την έγκριση της Washington να τον δολοφονήσουν και σε δύο εβδομάδες μετά δολοφονήθηκε και μετά επέλεξαν τον Ζωζεφ Καμπιλά και είπαν αυτός είναι νέος μπορούμε να τον ελέγξουμε είχε υπηκότητα Ρουάντας και θα μπορούσαμε να το κάνουμε πρόεδρο όλα αυτά λοιπόν είναι παρέμβαση αυτό που χρειάζεται το Κονγκό είναι να ξαναβρει την κυριαρχία του. Ένα στρατό που να μάχεται αποτελεσματικά. Μια μονοσκόπου να εξυπηρετεί τα συμφέροντα τη ειρήνη. Να σταματήσουν αυτοί οι αρπακτικοί ε, φορεί οι οποίοι συνδέονται με τις μεγάλες πολυεθνικές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στήρ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όπως αναφέρθηκε η σύραξη και η αστάθεια στο Κονγκό συσχετίζεται άμεσα με την μάχη για να κερδίσουν κάποιοι τα πολλά ορυκτά και μέταλλα που έχει αυτή η χώρα τον ορυκτό και μεταλλικό πλούτο που θα πρέπει από την άλλη πλευρά όμως να εμπλουτίζουν τους πολίτες ε, του Κονγκό. Είναι ωστόσο μια κατάρα για τη χώρα αυτή βλέπουμε τεράστιο ποσοστό των κατοίκων του Κονγκό ζει κάτω από το κατόφλι τη 43% των παιδιών πάσχει από μόνιμο υποσυτισμό. Θα ήθελα να συγχαρώ για αυτή την ε, ειρηνευτική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση ενός συστήματος υποχρεωτικού χαρακτήρα για τις εισαγωγές δίκαιες και τίμιε εισαγωγές βολφραμίου στην Ένωση που δεν θα προέρχονται από ζώνες σειράξεων στο Κονγκό και να σταματήσει πια αυτή η κατάσταση με τις σειράξεις και τους πολέμους για την εκμετάλλευση ορυκτών και ε, μετάλλων. Αλλά η μάχη για τα ορυκτά και τα μετάλλα δεν είναι το μόνο αίτιο, είναι και η διαφθορά, η έλλειψη χρηστής διακυβέρνησης και διαχείρισης. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να μην υπάρχει χειραγώγηση των προεδρικών εκλογών ε, του στο Κονγκό και να μην καθυστερήσουν υπερβολικά. Πιστεύω ε, ότι αυτό το πρόγραμμα για το Κονγκό, το 11ο αυτό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το κράτος δικαίου, τις μεταρρυθμίσεις ε, όσον αφορά τη δικαιοσύνη, την αστυνομία και το το στρατό και το ίδιο να ισχύει και για άλλα αφρικανικά κράτη, όπου η διαφθορά μπορεί να είναι μία από τις κυριότερες μάστιγες και ένα από τα κυριότερα αίτια των προβλημάτων, που ίσως όμως μπορεί να μην είναι τόσο προφανές όπως στην περίπτωση του Κονγκό. Αρένα παρακαλώ στη συνέχεια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά συζητάμε ένα ψήφισμα για τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Και όπως υπόθηκε δεν είναι η πρώτη και φοβάμαι πως δεν θα είναι η τελευταία. Σήμερα καταδικάζουμε τις φαγές στο Μπένι, που όπως είπε ο κύριος Πιτέλα, προστίθεται σε εκατομμύρια νεκρών στο Μπένι, πάνω από χίλια άτομα εσφάγησαν μέσα σε 1,5 χρόνο. Επίσης έχουμε απαγωγές, ε, καμένα σπίτια, βιασμούς, απειλές, οι πληθυσμοί που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους αυτή είναι η πραγματικότητα του κυβού. Όπως είπαμε, είναι αντικείμενο ιδιαίτερη επιθυμίας για το ε, χρυσό και το κολτράνιο αυτή η περιοχή. Πήραμε αποφάσει όμω για την ανεχνησιμότητα των ε, υλών αυτών, αλλά διστάσαμε να το κάνουμε. Και το Συμβούλιο δεν ήταν πάντα ιδιαίτερα θετικό έναντι των ετοιμάτων μας. Τώρα όλοι συμφωνούν ότι οι πολυεθνικέ μα πρέπει ε, να είναι πιο προσεκτικές για την κατάσταση της χώρας. Αλλά η αστάθεια που επικρατεί στη χώρα οφείλεται και στις αρχές της χώρας και είναι απαράδεκτη γιατί αφήνει εγκλήματα ατιμόρυτα. Και δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό. Πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες έρευνες εντός της χώρας και διεθνής για να εντοπιστούν οι υπέτειοι και για να υπάρξουν οι αναγκαίες ποινές. Επειδή είναι τώρα προεκλογική περίοδο, θα είναι δύσκολο, το ξέρουμε. Και τα εγκλήματα και οι παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι όλο και πιο πολύ άριθμα. Πρέπει λοιπόν ω Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεργαζόμενοι με την ε, Αφρικανική Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη, να συντονιστούμε ούτω ώστε να διεξαχθούν οι εκλογέ σε ειρηνικέ συνθήκε και διαφάνεια με σεβασμό του Συντάγματο. Όχι μόνο γιατί θέλουμε να γίνει σεβαστό το Σύνταγμα, αλλά γιατί είναι η μόνη εγγύηση για να επανέλθει η σταθερότητα, να αποφύγουμε τις κρίσεις που είναι ανθρωπιστικές και φυσικά να αποφύγουμε ο λαός που είναι το πρώτο θύμα να συνεχίσει να υποφέρει. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φωτίγκα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο λαός του Κονγκό θα πρέπει και πάλι ε, να υποστεί απίστευτες φρικαλαιότητες που προκαλούνται από τους παραστρατιωτικούς ή στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Είχαμε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας που βοήθησε σε αυτό. Ήταν η περίοδος της ε, μεταβίβασης της ε, εξουσίας. Θα πρέπει να τεθεί σε αυτο ηταν η περιοδος της μεταβιβασης της εξουσιας θα πρεπει να τεθει σε το νέο σύνταγμα το συντομότερο. Και θα πρέπει να αναλυθούν όσε συνέργειες χρειάζονται ε, με την εμπλοκή του διεθνού παράγοντα, ούτω ώστε να υλοποιηθεί η, το ψήφισμα αυτό του, του Μαρτίου και πω θα πρέπει να δοθεί ε, στην Μονούσκο η κατάλληλη εντολή και να μπορέσουμε να σταματήσουμε την ατιμορρησία και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα πρέπει να εμπλακεί και πάλι. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και στη συνέχεια, Βότμανς, 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κάνουμε λόγο εδώ και χρόνια για τον εμφύλιο πόλεμο στο Κονγκό και ξεχάσαμε πόσο όμορφη είναι αυτή η χώρα όταν είναι ειρηνική η κατάσταση που επικρατεί εκεί. Όμως τώρα σκοτώνονται άνθρωποι, δολοφονούνται άνθρωποι, γυναίκες ε, βιάζονται οι μητέρες ε, <clears throat> βλέπουμε ότι προτού οι ίδιες ε, δολοφονηθούν τα κορίτσια τους πέφτουν στα χέρια των ενόπλων της ε, Μονούσκο και οι γυναίκες βιάζονται κατά πλειοψηφία στο Κονγκό είναι μια μάστιγα αυτή αξιότιμοι συνάδελφοι όλα αυτά Ήδη πριν από 16 χρόνια τα γνώριζε επί που... η διεθνής κοινότητα. Μπορούν να μας εμπιστευτούν για ακόμα οι Κογκολέζοι μια και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και δεν αποκαθίσταται η ειρήνη και υπάρχουν τέτοιες τραυματικές εμπειρίες. Πρέπει να σκεφτούμε και τις επιπτώσεις όλων αυτών. Πρέπει να σκεφτούμε ότι το Κονγκό πάσχει, υφίσταται αυτά τα δεινά λόγω του φυσικού του πλούτου και ο Καμπίλα ε, έχει εκμεταλλευτεί αυτό το, αυτή την κατάσταση. Πρέπει να διασφαλιστούν όμως ελεύθερες, η διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Πρέπει να υποστηρίξουμε την ειρηνευτική διαδικασία με κάθε τρόπο και η εντολή του, της Μενούσκου πρέπει να πάψει η ατιμορρησία όσοι εγκλημάτισαν πρέπει να προσαχθούν στην δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν Πρέπει να υπάρξει μια προοπτική για τη δημοκρατία ώστε να έχει μέλλον. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια, Βερζιά, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η χώρα ζει μια δραματική κατάσταση. Όλο και περισσότερες άμπλες ομάδες, φτώχεια, αποσταθεροποίηση, σφαγές και αξιοποίηση των εθνοτικών διαφορών και αξιοποίηση των φυσικών πόρων από τις πολυεθνικές και τις γειτονικές χώρες, ιδιαίτερα της ευρωπαϊκέ. Τουλάχιστον 400.000 Κογκολέζοι είναι στην εξορία. 1,5 εκατομμύριο εσωτερικά μετατοπισμένοι. Πολλά εκατομμύρια νεκρών σε μια γενική αδιαφορία. Πρόκειται για γενοκτονία που το αναγνωρίζει από το 2010 ο ΙΕ. Είναι μία από, το πιο, από τις πιο μακροχρόνιες γενοκτονίες παρά την χαμηλή ένταση που είπε ο κ. Πιτέλα. Αλλά η βία τους τελευταίους μήνες αποδεικνύει ότι τίποτα δεν έχει καλυτερέψει. Πότε λοιπόν η διεθνής κοινότητα θα αντιδράσει. Οι ευθύνε είναι βαριέ. Διαφόρων. Ναι, πρέπει να σταθεροποιηθεί η χώρα και να καταλάβει ο κύριο Καμπιλά ότι πρέπει να δράσει λογικά. Βεβαίω πρέπει να γίνουν ανεξάρτητε έρευνε και για το ρόλο τη Μονούσκο. Πρέπει να μην χρηματοδοτούνται οι ένοπλε ομάδε και να μην πολλούνται τα ορυκτά του αίματο. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια η κυρία Ριβαζή, παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι θηριωδίες ε, συνεχίζονται στο Κονγκό. Το 2014 δώσαμε στον δόκτορα Μουκουέγγε το βραβείο Ζαχάροφ για τη δράση του για τα θύματα σεξουαλικής βίας. Αλλά σήμερα δεν είναι μόνο οι γυναίκες, ακόμη και τα παιδιά και τα μωρά εφίσταται τέτοιου τύπου ε, βία. Αξιοποιείται αυτή η σεξουαλική βία γιατί είναι όπλο μαζικής καταστροφής πέρυσι ο ΙΕ δημοσίευσε μια τρομερή έκθεση. να υπάρξουν νέοι μηχανισμοί για να σταματήσει η ασυδοσία. Είναι μια πρόοδο ότι μάθαμε ότι ορισμένοι δήμοι καταδικάστηκαν, αλλά δεν επαρκεί γιατί είναι συνένοχος και η κρατική εξουσία. Γιατί η βαρβαρία, η βαρβαρότητα αυτή έχει να κάνει με την έλλειψη κράτους στο Κονγκό και είναι κυρίως επίπτωση των παρανόμων εξορρυκτικών δραστηριοτήτων που προστατεύονται από τις ένοπλες ομάδες. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα για να καταπολεμήσουμε αυτά τα εγκλήματα. Διότι όλοι και όλες είμαστε υπεύθυνοι για αυτά τα αιματηρά ορυκτά που μπαίνουν μετά στα τηλέφωνά μας και τους υπολογιστέ. μας. Πρέπει κάτι να κάνουμε επιτέλους. Χάρη στην πρόσφατη συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ζέλα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν καλά μαντάτα για την Κεντρική Αφρική. Ο πρώην αντιπρόεδρος του Ζαν Πιέρ Μπέμπα λόγω εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας καταδικάστηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη μετά από εξαετή δίκη σε πολιετή φυλάξη. Αυτό κάπως αποκαθιστά τη δικαιοσύνη για τις γυναίκες, άνδρες και παιδιά που από τις στρατιωτικές του δυνάμεις δολοφονήθηκαν, ακροτηριάστηκαν, βιάστηκαν. Πέρα από αυτό όμως δεν έχουμε κάτι το θετικό να αναφέρουμε για την επίκαιρη κατάσταση στο Κονγκό. Έχει αυξηθεί πολιτική ένταση, η ένταση στη χώρα με κάθε τέχνασμα προσπαθεί ο πρόεδρος ε, Καμπιλά να παραμείνει στην εξουσία, να αναβάλει τις εκλογές, να παρατείνει με τεχνητό τρόπο την εξουσία του που θα τερματιζόταν κατά το έτος 2016. Υπάρχουν απαγορεύσεις ε, για διαδηλώσεις ε, της αντιπολίτευσης, πάλι νεκροί. Βλέπουμε εδώ ότι έχει ξεσπάσει μια κρίση που έχει οξύνει την ανθρωπιστική κρίση στη χώρα. Ιδιαίτερα πρέπει να εκφράσουμε τη θλίψη μας όμως ότι στην ανατολική περιοχή της χώρας συνεχίζονται οι σειράξεις με τους αποκαλούμενους επαναστάτες ε, και τις φρικαλαιότητες που προξενούν. Ε, κύριο αίτιο είναι η μάχη για να αποκτήσουν την πρόσβαση και τον έλεγχο στα ορυκτά και μέταλλα αυτής τη περιοχής ε, που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης στα ορυχεία εκεί. Υπάρχει εκτοπισμός, δολοφονίες, καταναγκαστική εργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο με τον νέο κανονισμό για αυτή την κατάσταση θα έπρεπε μέταλλα και ορυκτά να τα θέσει σε ειδική κατηγορία για τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να απαμβληθεί η κατάσταση. Δυστυχώς υπήρξε διαπραγμάτευση ένα κείμενο το οποίο ήταν γενικόλογο και αφηρημένο και έτσι, για παράδειγμα, τώρα θα παραμείνουν εκεί Αμερικανοί οι οποίοι θα υποτίθεται ότι ε, θα έχουν αποτέλεσμα για την απαγόρευση ή εξαγωγή αυτών των ε, ορυκτών και μεταλλευμάτων. Μπορούμε να λέμε ότι νομίζουμε ότι είναι σωστό, αλλά θα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο είναι σωστό στην πράξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Συν... Ε, και παρακαλώ. Σήμερα είμαι το Μπένιο γιατί σήμερα το πρωί δεν έκανα την καθημερινή μου διαδρομή, γιατί δεν κάθισα ήσυχη σπίτι με τα μωρά μου, γιατί δεν ζήτησα να έρθει μαζί ο σύζυγός μου, γιατί δεν αποφάσισα να είμαι με αυτούς, με τα 400 εκατομμύρια συμπατριώτες που άφησαν τη χώρα για να ξεφύγουν από τη βία, μα για να πάω πού, στην Ευρώπη, στην Νότια Αφρική. Και γιατί για να με στείλουν πίσω και να λένε ότι δεν δικαιούμαστε τη διεθνή προστασία. Και πού να γυρίσουμε στον Μπένι. Παρ' όλα αυτά, εδώ αισθάνομαι σίγουροι. Εδώ η έδρα του Μονούσκοβου είναι τόσο μακριά και αυτοί έχουν την εντολή να μας προστατεύσουν και έτσι η θελεδινής κοινότητα. Όμως είμαι μόνη μου. Έτσι η οικογένειά μου είναι σε ασφάλεια. Τουλάχιστον προς το παρόν και τους γλίτωσα αυτό το απάνθρωπο γιατί αυτά τα κτίνη δεν με ε, βίασαν απλώς αλλά με πλήγωσαν με μαχαίρια, με τσουγκράνες και μετά με κάψανε και ε, ακόμη είχα τις αισθήσεις μου αλλά δεν φοβόμουν και σκεφτόμουν εσάς, σκεφτόμουν τα παιδάκια μου και όλα που κράτησαν μόνο μια στιγμή. Παρ' όλα αυτά είμαι ε, πάρα πολύ χαρούμενη και αυτό ε, γιατί δεν κάθισα να, να δω στο χωριό αυτά τα οικεία πρόσωπα τα οποία θα έπρεπε να δουν αυτή τη σφαγή και αυτό γιατί στο τελευταίο μάντρωμα μας κάνανε ήμασταν κυρίως γυναίκες και, και, παιδιά βέβαια πάνω από πέντε ευτυχώ. Οπότε ξαφνικά τι είδαμε ότι δεν, δεν, δεν είδανε όλα, όλα αυτά τα σημάδια στο κορμί μου, αυτά τα, τα βασανιστήρια. Μετά από τις ώρες, ώρες που πέρασα στα βασανιστήρια και τελικά ε, ευτυχώς που η διεθνής ε, κοινότητα ενδιαφέρεται λίγο για αυτά που γίνονται εδώ στο ανατολικό μέρος της χώρας γιατί έχουν άλλα πράγματα να ασχοληθούν τα ΜΜΕ. Από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι το 2016 στον Μπένιτο και τον έχουμε 1.200 οι οποίε φαγιάστηκαν εν μέσω γενική αδιαφορία. Οπότε τώρα το κίνδυνο είναι η γενοκτονία. Ντροπή, ντροπή. Όχι την ατιμορρησία. Πότε θα έρθει η δικαιοσύνη. Σα ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ Στη συνέχεια σας ευχαριστούμε και για το ότι ε, μιλήσατε στην ε, αρχική γνώση και στη συνέχεια Τσαρνέτσκι παρακαλώ. Ε, e, σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τον λόγο. Η προλαλή σας προέρχεται από την Ιταλία και όσα πρέπει να γίνουν είναι ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε αυτό το ψήφισμα να αποκτήσει σάρκα και ωστά. Δεν επαρκεί πρέπει να πούμε ότι ψηφίσματα επί θα εγκρίνονται ψηφίσματα που προσυπογράφουν όλοι παντού στον κόσμο, αλλά να μην γίνεται τίποτα. Δεν επαρκεί αυτό. Πρέπει κάτι να πράξουμε ώστε το ποινικό δίκαιο να χρησιμοποιήσουμε ώστε να πετύχουμε κάτι. Να προσαχθούν σε δικαστήρια εκείνοι που είναι ένοχοι και έχουν διαπράξει εγκλήματα. Η Ευρώπη δεν, δεν μπορεί να τηρήσει εισηγήν ισχύω. Πρόκειται για την ίδια την τιμή και την αξιοπρέπειά μα. Και οφείλουμε σε σχέση με τι χώρε που κάποτε ήταν δικές μας απικίες να δράσουμε με αυτόν τον αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Διάστε μέρα παρακαλώ. Δύο λεπτά. Η δημοκρατία του Κονγκό αντιμετωπίζει μια ανθρωπιστική κρίση που είναι η μακρύτερη της ιστορίας του. Οι σφαγές και οι επιθέσεις ε, στην ανατολική περιοχή έχουν δημιουργήσει πάνω από 13 εκατομμύρια εσωτερικά μετατοπισμένων και μισό εκατομμύριο εξορισμένων. Γίνονται επιθέσεις, σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες και παιδιά, χίλιοι βιασμοί τη μέρα, επιθέσεις αδιάκριτες και στρατολόγηση παιδιών για μαχητές. Είναι τρομερές αυτές οι ενέργειες των Μπένι, τον Λουτέρα και των Μπουτέμπο ε, είχαν ως αποτέλεσμα χίλιες δολοφονίες. Εκφράζω την αλληλεγγύη μου και τη στήριξή μου στα θύματα και τις οικογένειές τους. Θα ήθελα να επιμείνω στην ανάγκη να ξεκινήσουν οι κοινέ επιχειρήσεις μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και της Μονούσκο. Είναι η μόνη δυνατότητα, κατά τη γνώμη μου, να αντιμετωπιστούν οι άθλιες ενέργειες των ένοπλων ομάδων όπως ε, των δυνάμεων της Ρουάντα ή άλλων δυνάμεων. Επιπλέον, οι αρχές της χώρας πρέπει να αντιμετωπίσουν τάχιστα την παράνομη εξόριξη ίδιων πόρων όπως το βολφράμιο, το τουξτένιο και το κασίτερο για να κλείσουν οι στρόφιγγες χρηματοδότησης των ενόπλων ομάδων. Επιπλέον, υπάρχει αναγκαιότητα να διεξαχθούν οι επόμενες προεδρικές εκλογές και οι κοινοβουλευτικέ. Θα ήταν αποτελεσματικό κάτι τέτοιο για να επανέλθει η σταθερότητα και η πρόοδο. Πρέπει η χώρα να αποκτήσει θεσμού τάχιστα. Πρέπει να μεταρρυθμιστεί η πολιτική και η στρατιωτική δικαιοσύνη για να σταματήσει η ατιμορρησία και να προστατευτούν οι πολίτε. Οι καταδίκες, η καταδίκη του Μέμπα από το δικαστήριο της Χάγης πρέπει να παίξει ρόλο παραδείγματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια ο κύριος Παντσέρη. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση στο Ανατολικό Κονγκό είναι αρκετά ξεκαθαρή και η ανταπόκρισή μας δεν έφερε αποτελέσματα μέχρι σήμερα γιατί νομίζω ότι πρόκειται για κροκοδίλια δάκρυα αυτά που έχουν χυθεί στο ημικύκλιο. Γιατί στο Συμβούλιο δεν πέρασε ο κανονισμός σε σχέση με τους ε, πόρους που παράγονται στην περιοχή, μέταλλα κλπ. Τι έκανε το Συμβούλιο και η Επιτροπή έδειξαν υποκρισία και σχιζοφρένεια. Θα έπρεπε να έχουμε μια ελάχιστη συνέπεια σε σχέση με τα όσα λέμε. Τα πράγματα είναι σαφή κάποια σημεία θα έπρεπε να ξεκαθαριστούν, να υπάρχει ενιαία πλατφόρμα και να μην δείχνουμε προς όλα τα μέτωπα αυτήν την ανικανότητα. Ο πρόεδρος Καμπίλα θα πρέπει να φύγει, να υπάρξει μετασχηματισμός πολιτικός. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι ανεπαρκής η λειτουργία του τακτικού στρατού θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι και ο ΙΕ είναι ανεπαρκής στις επιτόπου επιχειρήσεις. Δεν έχουμε μπορέσει να θέσουμε ένα φρένο, ένα τέρμα σε αυτή την κρίση. Η Ουγγάντα και η Ρουάντα δεν κάνουν τίποτα ενώ έχουν εμπλακεί το αντίθετο. Άρα χρειάζεται να συγκροτηθεί μια διεθνής επιτροπή, μια έρευνα του ΟΗΕ, ούτως ώστε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε τάξει. Θα πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Να βγει η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτή τη φάση της ανικανότητας και ανικανότητας λήψης αποφάσεων. Ο κύριος Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Κούκαν, 1,5 λεπτό παρακαλώ. The DRC lives in a... Ευχαριστώ. Η χώρα αυτή ζει σε μια κατάσταση τεχνητής ειρήνης και τεχνητής ασφάλειας. Η τελευταία έκρηξη βίας ε, στο βόρειο τμήμα της χώρας δημιούργησε άθλια εντύπωση εκατοντάδες δολοφονιών, εξαφανίσεις, βιασμοί και καταστροφή ζωτικών υποδομών. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι η διεθνής αντίδραση ήταν ε, πολύ περιορισμένη και ανεπαρκής. Οπότε, πρώτο στόχος είναι να σταματήσει η βία και όλες οι ενοπλές ομάδες πρέπει να καταθέσουν τα όπλα τους. Η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένη και τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδείξουν περισσότερη παρουσία, να είναι πιο κατηγορηματικές, να παίξουν περισσότερο ρόλο, να δώσουν στήριξη στην προσπάθεια αφοπλισμού. Η Μονούσκο πρέπει να έχει δυνατότητα να αντιδρά ταχύτερα για να προστατεύει τον ε, άμαχο πληθυσμό. Επιπλέον πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες για τα εγκλήματα και να διωχθούν οι υπεύθυνοι. Εάν δεν ε, τιμωρηθούν οι πέτοι, αυτή η ατμόσφαιρα τιμωρησίας θα συνεχίσει να δηλητηριάζει το κλίμα και μπορούμε να περιμένουμε και περαιτέρω εκρήξεις βίας. Είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες της χώρας αξίζουν μια καλύτερη μοίρα μετά από 20 χρόνια συγκρούσεων και βίας. Ευχαριστώ πολύ, λέει πρόεδρος. Ο κύριος Φουντσούλικα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ανησυχώ πάρα πολύ γιατί η κατάσταση επιδρώνεται συνέχεια στο βορειοανατολικό Κονγκό. Και έχουμε ένα σωρό μαντάτα που έρχονται για αυτή την υποχρεωτική ε, στάτολόγηση ανηλίκων για την ε, βία και θα πρέπει να απευθυνθούμε στην κυβέρνηση και στην Μονοσκό ώστε να γίνει κάποια έρευνα για να δούμε ακριβώς για να εξάρτητοι να αποδώσουν τις ευθύνες για τα λάθη της κυβέρνησης και της Μονοσκό. Θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να ασχοληθεί με αυτές τις σφαγές και να δούμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Δεν υπάρχει αποτελεσματικός στρατός ε, να υπάρξει ασφάλεια σε μπαίνει λουμπέρο και μπορεί να, να προστατεύσουν τον κόσμο. Θα πρέπει να δούμε το πώ θα σταματήσουν τα σεξουαλικά εγκλήματα, σεξουαλική βία. Οι υπεύθυνοι να προσαχθούν ενώπιον τη δικαιοσύνη και ενώπιον του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου. Πρόεδρο, σε ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Ο κύριο Σασί, ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τι τελευταίε δεκαετίε η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό ήταν το σκηνικό της ε, προαγωγή τη Βία που στήχησε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπου. Το σενάριο είναι πολύ ανησυχητικό. Πρόσφατα μια ομάδα πραγματογνωμόνων ε, είπε ότι ένα παρόμοιο σενάριο μπορούσε να διεξαχθεί σε σχέση με τον Μπουρούντι με την αντιπαράθεση πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για τις προεδρικές εκλογές 2017 κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί δυστυχώς. Τώρα φτάνουν μαντάτα ειδήσει για σφαγέ σε σχέση με ε, ενόπλους στην νοτιοανατολική περιοχή της χώρας. Δεδομένου όλων αυτών πρέπει να πράξει ό,τι περνάει από το χέρι τη η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην κλιμακωθεί η κατάσταση. Σε σχέση με τα όσα συνέβησαν το 1994 στη Ρουάντα, καθώ επίση και με του δύο εξοντοτικού πολέμου του Κονγκό, πρέπει να τα θυμόμαστε όλα αυτά για να δράσουμε άμεσα αποτελεσματικά. Έχει παράσχει βοήθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση τη φτώχεια και την αποκατάσταση των πραγμάτων στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παράσχει τη βοήθειά τη ώστε να κληθούν οι ε, κογκολεζικέ αρχέ να σεβαστούν τα δικαιώματα Τη της και του ανθρώπου και να μπορέσει ο διάλογος να προαθεί σε σχέση με την Αφρικανική Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάιερ. Ευχαριστώ. Έξι εκατομμύρια χρόνια, ε, νεκροί τα τελευταία χρόνια. Αυτό αποδεικνύει ότι η καταπολέμηση τη περιφερειακή τρομοκρατία αλλά και τη Ισλαμικής τρομοκρατία σε αυτή την περιοχή, η καταπολέμηση του Μπόκο Χαράμ και του Σαμπάπ δεν έχει επιτύχει η έξοδος από την Σομαλία σε όλη την υπόλοιπη Δυτική Αφρική της τρομοκρατίας είναι πραγματικότητα. Δεν ε, πετυχαίνουμε και πολλά με τις προσπαθίες μας. Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει απλώς να λέει μεγάλα λόγια. Πρέπει να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε ότι θα συνεχιστεί η κατάσταση μέχρι ότου το κολτάνιο και άλλες πρώτες ύλε να μην αξιοποιούνται από αυτές τις ένοπλες ομάδες και να μην πολλούνται στις δικές μας εταιρείε. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε τις αναγκαίες ενέργειες. Πολλά λέμε σήμερα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. Γιατί φαίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να θίξουμε την κατασκευή τηλεφώνων, κινητών. Σα Σας ευχαριστούμε. Σημαντικό είναι να εκφράζονται οι απόψει μα. Ολοκληρώσαμε τώρα τι παρεμβάσει αυτές. Ακολουθεί το Catch the Eye. Ο πίνακα είναι πολύ σύντομος. Ο κύριος Καπούτο παρακαλώ πρώτος. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ασχολούμαστε για τρίτη φορά στο Κόγκο. Η κατάσταση είναι τραγική στη χώρα και πάρα πολύ πρόσφατα ανακαλύψαμε ε, εκατοντάδε πτώματα ε, σε γίνους ε, τάφου, Το έγινε το 2014 και με ματσέτες είχαν σφαγιάσει γυναίκες και παιδιά. μετά κάθε λεπτό μία γυναίκα βιάζεται. Έχουμε πάνω από 1.500 οι οποίοι έχουν απαχθεί κάθε μέρα. Και έχουμε τώρα αυτή ε, στις συμμορίες των ενόπλων που προβαίνουν σε γενοκτονία και ζητείται επομένως κάποια έρευνα για όσα γίνονται στο βόρειο Κιβού. Θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ρόλος της Ρουάντα. Χρειάζεται τώρα περισσότερο από ποτέ να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνείς να τα σταματήσουν αυτές οι σφαγές. Θα πρέπει να δούμε πώς θα βοηθήσουν οι οργανώσεις που δουν τόπου, ο ΟΗΕ, να γίνει αυτή η διεθνής έρευνα του ώστε να σταματήσει η τραγωδία. Κύριε Μαριά, το λόγο. Πρόεδρε, η λαϊκή δημοκρατία του Κογκό είναι η μεγαλύτερη χώρα της κεντρικής Αφρικής και συνάμα μια από τις πλουσιότερες σε ορυκτά. Δυστυχώς όμως εκεί οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και η έξαρση βίας που γνωρίζει η χώρα αυτή. Τον περασμένο Δεκέμβριο υπερψηφίσαμε πρόταση που καταδίκαζε τις παράνομες δραστηριότητες εξόριξης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Εθνικό Πάρκο Βιρούγκα, ένα πάρκο με τη μεγαλύτερη βιοπικιλότητα στην Αφρική και παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO οι βεοπραγίες στην περιοχή του βόρειου κίβου ξεκινάνε περίπου την ίδια περίοδο που διεξάγονται οι πρώτες σεισμολογικές έρευνες στο τέλος του 2014. Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα μετράμε ήδη περισσότερους από 600 νεκρούς. Αποτρόπιες σφαγές στην περιοχή Μπένι το Μάιο, με θύματα εγγύους, μικρά παιδιά και ηλικιωμένους η ευρωπαϊκή ένωση οφείλει όχι μόνο να καταδικάσει αυτές τις απάνθρωπες πράξεις αλλά και να λάβει αυστηρά μέτρα για να σταματήσει οποιαδήποτε ανάμειξη ευρωπαϊκών πολιεθνικών στι παράνομε δραστηριότητε που λαμβάνουν χώρα στο ανατολικό κονγκό. ιδιαίτερα πρέπει να εξετάσει τι καταγγελίε συνεργασία πολιεθνικών εταιριών με ομάδε ενόπλων με στόχο την τρομοκράτηση και τον διωγμό των ντόπιων πληθυσμών. ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάκοφτσιτς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς η RDC, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είναι σήμερα ένα από τα υποδείγματα για το ότι ο πλούτος μπορεί να μετατραπεί σε μια κατάρα, σε μάστιγα. Κυρίως όταν ο πλούτος δεν φτάνει στους πολίτες μιας χώρας, αλλά παραμένει στους θύλακες των πολιτικών ελίτ, στις τσέπες των προνομιούχων. Και για αυτούς τους λόγους θα ήθελα να σας προτείνω ότι στην περίπτωση αυτή τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό πρέπει να δράσουμε διτά, με δύο τρόπου. Αληθεύει ότι είναι το τρίτο ψήφισμα για το οποίο κάνουμε λόγο, με κάποια μεν αποτελέσματα, όμω πρέπει να καταφέρουμε να πετύχουμε πρώτον το ποινικό δικαστήριο τη Χάγη να τοποθετηθεί με κάθε σαφήνεια όπω έγινε πρόσφατα. Διότι αυτή είναι μία οδό ώστε να εξευρεθεί μια ειρηνική λύση και γνωρίζω από την ίδια την πείρα από την πρώην Ιουγκοσλαβία όπου υπήρξαν τέτοιες σειράξεις και τερματίστηκαν μέσω του ποινικού δικαστηρίου της Χάγης. Θα πρέπει στη συνέχεια να υποστούν κυρώσεις οι πολυεθνικές, κυρίως οι ευρωπαϊκές, που συνεχίζουν να παραβιάζουν τα δικαιώματα τα οποία εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε. Δηλαδή, πρέπει να αποφύγουμε να χρησιμοποιούνται ορυκτά και μέταλλα, φυσικός πλούτος της περιοχής αυτής για να ανατροφοδοτείται η σύραξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα φτάσαμε στο τέλος. Ο κύριος Ναύρατσης θα πάρει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψε και γι' αυτό ευχαριστώ του βουλευτέ που ήταν ξεκάθαρε τοποθετήσει του Ορισμένοι εκ των αξιωτήμων ε, βουλευτών πάντω δεν είπαν για τι συνέπειε των μέτρων μα και του ψησματό σα Το Πώς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε στο Συμβούλιο Εξωτερικών στις 23 Πέμπτου κάποια συμπεράσματα που αφορούν την δημοκρατία του Κονγκό και που συγκλίνουν ως το κείμενο της 10 Μαρτίου του ΟΗΕ. Και μιλήσαμε για την ευθύνη, για την δικαιοσύνη και την ασφάλεια στη χώρα. Επίσης, τα σημερινά 23 Μαΐου είπαμε ότι θα πρέπει κάτι να γίνει για αυτή την κατάσταση και ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε ε, όλα τα μέσα που έχουμε στην διάθεσή μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους για το ότι έχουμε 7 κείμενα προτάσεων ψηφισμάτων που έτσι